την προσπάθειά μας να δώσουμε ένα μέλλον, μια προοπτική για το μέλλον στους πολίτες του Ιράν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βέλτερ. Κλείνει αυτό το θέμα. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης, για την 16η τη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη. Έχει το λόγο η Λέβη Άστον. Uh, Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία σήμερα το απόγευμα να συζητήσουμε και για το έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποτελέσματά του. Δηλαδή. Όπως ξέρετε μίλησα σε αυτό το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα μαζί με πολλούς υπουργούς εξωτερικών από όλο τον κόσμο. Με εκείνη, ε, ε, με εκείνη την ευκαιρία βεβαίως η Λιβύη ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Χαίρομαι που η παγκόσμια κοινωνία έδωσε ένα έντονο μήνυμα όσον αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη. του ε, Ήδη άλλωστε είχε προταθεί η αναστολή ε, της ιδιότητας τους μέλους για τη Λιβύη και αυτό επιβεβαιώθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΓΕ. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι πολυμερείς οργανισμοί μπορεί να ανταποκριθούν στην εντολή τους και μπορούν να ενεργήσουν και επίκαιρα, άμεσα, εγκαίρως. Το Συμβούλιο αυτό έχει την ευθύνη οι δηλωμένες προθέσεις να μετατρέπονται σε πραγματική δράση και πρόοδο. Νομίζω ότι η κυρία Πιλέη, η πατή ε, αρμοστής στη Γενέβη δίνει τη σωστή κατεύθυνση πολιτικά ακριβώς ώστε να είναι διαφορετικά τα πράγματα στην πραγματικότητα. Ε, σημασία δεν έχει ο αριθμός των ψηφισμάτων αλλά πώς αντανακλώνται αυτά ε, στην πραγματική ζωή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακούμε ότι ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εξαγάγει ευρωπαϊκές αξίες σε άλλους. Η ισότητα και η δικαιοσύνη δεν είναι ευρωπαϊκά δικαιώματα, είναι παγκόσμια και ποτέ δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να πιστέψουμε ότι άλλοι άνθρωποι στην Αφρική, στην Ασία ή οπουδήποτε ε, πρέπει να προασπίσουν λιγότερο τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό υπεραμεινόμεθα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοποθετούμεθα κατά των παραβιάσεων. Όπου και αν συμβαίνουν, η προστασία δεν υπήρξε πάντοτε ευθεία γραμμή. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες και στην Ευρώπη. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζητά προκλήσεις, ανταλλάσσει εμπειρίες και βοηθά αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Είχαμε πολλές προτεραιότητες για την 16η Σύνοδο και τις συζητήσαμε ενεργά με τους εταίρους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε μια πρωτοβουλία για την ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, του δόγματος κατάργηση της βίας σε διάφορα μέρη του κόσμου για θρησκευτικούς λόγους. Ταχθήκαμε λοιπόν υπέρ της ελευθερίας, της λατρείας, του δόγματος και της θρησκείας. Παντού. Επίσης υποβάλαμε ψηφίσματα για τη Βούρμα, Μιανμάρ και για την Κορέα, τη Λαϊκή Δημοκρατία. Πιστεύουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό χρειάζεται ειδικό συζήτης. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την δημιουργία ενός ειδικού ε, εισηγητή, εισηγητή για το Ιράν, δηλαδή ανησυχούμε σοβαρά για την υποβάθμιση της κατάστασης στο Ιράν. Και αυτό τονίστηκε και από την κυρία Ναβί Πιλέ. Ανησυχούμε ακόμη με τον αριθμό των θανατικών καταδικών πάνω από 100 φέτος, όπως είπαμε ήδη στην προηγούμενη συζήτηση. Και έχουμε καταπίεση όλων αυτών που θέλουν ελευθερία του λόγου και του συναθρίζεστε. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα άμεσα και σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει την πρόσκληση της Αιγύπτου προς την κυρία Πιλέ να στείλει στελέχη της στην Αίγυπτο Πιστεύουμε ότι θα ε, υλοποιηθεί η αποστολή του ταχύτερο δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης μαζί με τις αρχές της Τινησίας θα υποβάλει ψήφισμα για την προώθηση της τεχνικής αρρωγής και βοήθειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μεταβατικές περιόδους. Επίσης υπάρχουν και άλλες ε, σοβαρές καταστάσεις όπως η Λευκορωσία και οι πολιτικοί φυλακισμένοι, το Κονγκό, όπου υπάρχουν συνεχείς εκθέσεις παραβιάσεων, ειδικότερα δεν υπάρχει σεξουαλική βία στο Κονγκό, καθώς και στην Côte στην ακτή του Ελεφαντοστού. Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συζητήσει, οι συγητέ, τα ψηφίσματα, αλλά όλα αυτά είναι το κομμάτι της εισρωή. Το θέμα είναι τι έκροε θα έχουμε για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε μια διαφορά επιτόπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αγωνιστεί να ενισχύσει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει ειδικότερα επίγουσες καταστάσεις. Και αυτό είναι βασικός στόχο μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Θα πιέσουμε για να έχουμε φιλόδοξο αποτέλεσμα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Άστον. Περνάμε τώρα στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, η κυρία Αντρίκενε έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, συνάδελφοι, θα ήθελα να υποστηρίξω πλήρως την απόφαση της, 1ης Μαρτίου του, των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την απόσυρση του Καντάφη από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην έκθεσή μου ως προς το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών μίλησα για τα κριτήρια συμμετοχής στην ε, κοινοβουλευτική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ελήφθηκαν πολύ σωστές αποφάσεις Μιλώντας για τη 16η Σύνοδο θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σε αυτή τη διαδικασία τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να ενισχύσει τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια αυτά. Και πιστεύω ότι αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να είναι πολύ ε, σωστή και συμπεριληπτική, να λάβουμε υπόψη τις μη κυβερνητικές και την κοινωνία των πολιτών. Τέλος, Βαρόνι Άστον, θα ήθελα να καλωσορίσω το Διευθυντήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας στο, στη δική μας ΚΕΠΑ. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να διοχετεύσουμε τη δράση μας προς την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, έτσι ώστε να υπάρχει καλός συντονισμός προσπαθειών, έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και ενωμένοι πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν από τους σοσιαλιστές για δύο λεπτά το λόγο έχει, το λόγο έχει ο κύριος Χάουιτ. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω την, ε, τον διορισμό της κυρίας Ζάρες ε, στην ε, Γενέβη για θέματα ε, ισότητας των φύλων. Καλωσορίζουμε την διορισμό της. θα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή γιατί η παγκόσμια, ο παγκόσμιος σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων με ειδικέ διαδικασίες και ο η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν ε, βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος που προσπαθούμε να προασπιστούμε. Είμαι απογοητευμένος που το έγγραφο που προέκυψε δεν αναφέρει ειδικέ συνεδριασίε, δεν υπάρχουν απαιτήσει για τα κράτη-μέλη να δικαιολογήσουν την άρνηση των χωρών να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες αξιώσει και δεν αναφέρεται και καθόλου σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Είναι ηρωνικό το γεγονός ότι μιλάμε για 7 χώρες για τη Λιβύη και για την ακτή του Λεφαντοστού μεταξύ αυτών. Θα πρέπει να βρούμε τρόπος να διασφαλίσουμε ότι όσοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να τιμωρούνται. Θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις στην υπατή εκπρόσωπο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη, δημοκρατική, τη δημοκρατία του Κονγκό, θα υποστηρίξουμε την ε, ε, διορισμό ειδικού εντεταλμένου για τη χώρα αυτή. Κατά δεύτερον, αποδέχεστε ότι σε κάποιο σημείο θα πρέπει να κρίνουμε για το κατά πόσον οι Παλαιστινιακές και Ισραηλινές έρευνες πληρούν τα διεθνή πρότυπα σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη αναφορά και στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο σε περίπτωση που δεν τα πληρούν. Και τρίτον, θα υπάρξουν ενστάσει σε ό,τι αφορά το Πακιστάν και το άρθρο 40 και την υποχρέωση αναφορά για πολιτικά και ε, μη δικαιώματα. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι παραβιάζεται, ότι αναστέλλεται η συμμετοχή της Λιβύης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, θεωρώ ότι είναι ε, χωρίς προηγούμενο. Εξονόντως των φιλελευθέρων για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις επίγουσε καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, στο Ιράν, στη Βερμανία, στη Λιβύη, την Ισία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά και οριζόντια θέματα τα οποία αφορούν τη βία, το βιασμό, ε, την προάσπιση της ελευθερίας. Δηλαδή το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λειτουργήσει σφαιρικά. Αλλά δεν έχει αξιοπιστία. Έχει διπλά πρότυπα και μέτρα και σταθμά και δεν μπορεί να ενεργήσει αρκετά γρήγορα. Όπως και η ΕΕ. Μέχρι σήμερα η ΕΕ δεν θέλησε να μελετήσει πραγματικά την απόδοσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είτε πρόκειται για απελάσεις, για εκδόσεις ε, ή την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Η Λιβύη ήταν μέχρι προχθές μέλος του ΟΗΕ και χαιρόμαστε που τέλος πάντων σταμάτησε να είναι. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος των Πρασίνων για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με άμεση δράση κατά της Λιβύης το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ απέδειξε ότι μπορεί να ενεργήσει όταν απαιτείται, μπορεί να ενεργοποιηθεί, μπορεί να... Ε, απέδειξε μάλλον ότι διάφορες περιφερειακές ομάδες συνενώθηκαν και το Συμβούλιο δεν χρειάζεται να είναι διχασμένο. Σήμερα δεν υπάρχει πια λόγος γιατί η δράση ε, για το Ιράν, για τη Βερμανία, για το Σουδάν, για ε, την Κορέα δεν πρέπει η δράση αυτή να ακολουθήσει ε, η εποχή μας είναι σημαντική και για άλλο λόγο. Έχουμε πρώτη λεπτομερή αναθεώρηση του, του έργου του Συμβουλίου και των ρυθμισεών του. Λυπάμαι που το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να καταλάβει τη σπουδαιότητα Τη αναθεώρηση αυτής. Ε, τουλάχιστον όμως η ανεξαρτησία του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των ειδικών διαδικασιών δεν υπονομεύθηκε και πρέπει να πω ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες αυτό είναι ήδη επίτευμα. Μελλοντικά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα πρέπει να δημιουργήσει συμμαχίες και να συνενωθεί με άλλους εταίρους. Θα πρέπει να ακούει και να συμβιβάζεται. Νομίζω ότι είχαμε πολύ καλή συμμετοχή από τον ύπατο εκπρόσωπο πριν από μερικές εβδομάδες και χαίρομαι που κάνατε αυτό το βήμα κυρία Άστον και κάνατε μια τόσο καλή παρουσίαση. Τελευταίο σχόλιο. Η απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της δημιουργίας της σχετικής διεύθυνσης στην υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων η, αντιπρο... αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενέβη θα παίξει σημαντικό ρόλο. Χρειάζεται ενισχυμένους πόρους και το έργο της πρέπει να ενταχθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης. Χαίρομαι που είμαι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη 16η Σύνοδο. της το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Άστον, χτες μέσα στα πλαίσια αυτών των κλειδονισμών και ανακατατάξεων resultado de una apuesta de desregular el mercado y la verdad es que usted tiene una gran dificultad precisamente porque esa orientación de fondo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 και να λάβουμε υπόψη την πολιτική γειτονίας η οποία μας οδήγησε σε μία βαθύτερη σκέψη ως προς τις εξελίξεις και στη Βόρειο Αφρική. Μιλάμε για την εξωτερική μας πολιτική, για το ελεύθερο εμπόριο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 2 των συνθήκων σύνδεσης ούτε με την Τίνιδα, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με τον ε, Νετανιάχου. Και επίσης θα μην μας πείραζε το ότι θα έπρεπε αυστηρά να τηρηθούν οι ρήτρε για ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά αυτή τη συμφωνία σύνδεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εκκρεμεί και οπότε και γι' αυτό ελπίζω ότι τελικά εδώ πέρα θα περάσει αυτό το κείμενο όπω πρέπει. Ευχαριστώ κύριε Μάγκερ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα για την Ευρώπη Ελευθερία και Δημοκρατία, για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Σαλαβράκο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κυρία Άστον, δεν θα πω ότι οι άνθρωποι είμαστε υποκριτές θα πω όμως ότι είμαστε αντιφατικοί. όλη η παγκόσμια φιλοσοφία όλη η λογοτεχνία όλοι οι λόγοι και εμείς όλοι σε αυτή την αίθουσα αναγνωρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και όμως όπως είπατε εσείς στις μισές χώρες μέλη του οηε παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. κάνουμε μια ραψοδία όχι ουσία. εν ονόματι μεγάλων ιδεών ξέρουμε ότι έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ανθρωπότητα με την έννοια αυτή χαιρετίζω την 16 έκτη σύνοδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη γενέβη και ελπίζω στην εποχή που εξελίσσεται και με τα διδάγματα της πείρας που έχουμε να λάβει ουσιαστικές αποφάσεις. ξέρετε έχω 40 χρόνια δικηγορία και έχω αντιληφθεί και έχω ως πίστη μου το γεγονός ότι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στάση ζωής. δεν επιβάλλεται εύκολα σας παρακαλώ κάντε ουσιαστικότερη πολιτική πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, προς τον κύριο Σαλαβράκο. Και τώρα, η επόμενη ομιλητές για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Βάιντερ. Κύριε Πρόεδρε. Κυρία Στον. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια πλατφόρμα διεθνή. Συγκροτήθηκε για να προαγάγει ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία παντού, σε όλο τον κόσμο. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχει διαδραματίσει και νομίζω ότι το Συμβούλιο έχει κάνει πάρα πολλά επένετα, όπω και βοήθεια προ την Αίγυπτο και για τη Λιβύη. Παρ' όλα αυτά όμω, ε, πολλέ φορέ δεν έχει την αφοριστικότητα, δεν ενεργεί ε, έγκαιρα, ε, δεν υλοποιεί τους στόχους, δεν υπάρχει ούτε καν διαφάνεια για στο το Συμβουλίο, δεν ενεργοποίησε κάποιους μηχανισμούς ε, επιχειρησιακούς και δεν μπόρεσε παλαιά προβλήματα να αντιμετωπίσει, όπως το στο Ιράν. Όμως, διακόπτει ο Πρόεδρος, σας παρακαλούμε. Μήπως μπορείτε να μιλήσετε λίγο βραδύτερα, λέει ο πρόεδρο, διότι είναι αδύνατο να μεταφραστείτε λόγω της τόσης ευγλωτία σας. Συνεχίζει ο μιλήτρια στον ίδιο ρυθμό. Τα, τα μέλη του Συμβουλίου, επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουν έναν δυναμικό διάλογο και κατά τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των συνόδων και θα πρέπει να υπάρχει επαφή με τις ομάδες και ε, προσοχή οι κακές πρακτικές να μην οδηγούν σε επιλεκτικές συζητήσεις για κάποια ζητήματα και έτσι να υπονομεύουν το κύρος του το ίδιο. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ένα διάλογο πιο ζωντανό με την κοινωνία των πολιτών απλά στο Συμβουλίο. Αλλά και μέσα και με κυβερνήσει οργανώσει. Κατά τρίτο λόγο, επίση, θα πρέπει να σα τονίσω ότι χρειάζεται να μπορέσουμε να αναλάβουμε πιο δυναμικό ρόλο ή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και εκεί θα πρέπει να ακούγεται ενιαία η φωνή τη ε, κοινότητα. Ε, θα, νομίζω ότι έτσι θα πρέπει εσείς ε, ε κυρία Υπάτη εκπρόσωπη να μας εκπροσωπείτε και επομένως θα πρέπει να συνοηθείτε με την Υποεπιτροπή των Δικαιωμάτων όσον αφορά την υποκαιρμοστία. Τώρα, επομένω, αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για το Συμβούλιο. Ότι θα πρέπει να προωθήσει και να βοηθήσει όλε αυτέ τι δημοκρατικέ αλλαγέ στην Μέση Ανατολή. Και επίση έχουν προσπαθήσει να φρενάρουμε το, το, το, το, το ριζοσπαστισμό, γιατί είναι κάτι το οποίο δυναμητίζει την διεθνή ασφάλεια. Και για αυτό σα λέω ότι η αποστολή ή στην Αίγυπτο θα ακολουθηθεί από άλλες αποστολέ στη Μέση Ανατολή ε, σε, σε ακόμα πιο επιθετικό περιβάλλον και ακόμα πιο περίπλοκο background και ατμόσφαιρα. σα ευχαριστούμε λοιπόν και τώρα για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισοτιμία για μας όλους είναι πολύ σημαντικότερο από το να επιτρέπουμε να παίζονται παιχνίδια, ε, να υπάρχει παιχνίδι εξουσίας και ίσως ε, και τα εμπορικά συμφέροντα να προηγούνται αυτών των τόσο σημαντικών αξιών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αντιμετωπίζεται από τη διεθνή κοινότητα απόλυτα στοχευμένα. Νομίζω ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Είδαμε ότι στην, ε, η αποστολή στην ε, την Ισία τα κατάφερε και αυτή στην Αίγυπτο και τώρα η Λιβύη. Η Λιβύη έχασε την θέση της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι σημαντικό, μια σημαντική απόφαση για να δείξουμε ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η κατάσταση, αλλά βέβαια συμβαίνει επίσης αποστολές, ε, ψηφίσματα και ίσως ε, και άλλα παρεμφερή θέματα ε, δεν επιτυγχάνουν. Γιατί έχετε δίκιο κυρία Αστον ότι δεν χρειάζεται να αποφασίζει κανεί κάτι, πρέπει να καταδεικνύει και τον δρόμο. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, συμβάλλει περισσότερο ε, στο μέλλον από ό,τι αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν σημαντικό τα Ηνωμένα Έθνη να δεχθούν ότι η κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα είναι διαφορετική από ό,τι πριν από αυτή. Και θέλω να σα καλέσω κυρία Υπατή εκπρόσωπε έτσι έτσι ώστε κυρίως εκείνοι οι οποίοι ανέκαθεν έλεγαν ότι είναι φίλοι μας, εκείνοι που εμείς ε, τους ε, θεωρούσαμε φίλους μας, ε, ειδικά αυτοί στο μέλλον να μην ξεχνάνε ότι είναι φίλοι μας και όχι όπως συνέβη αυτό με την ψηφορία το Σεπτέμβριο όπου αφήσανε στα κρύα του Λουτρού την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ένα λεπτό το λόγο ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή τη συζήτηση και πάλι θα τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Έχει σβήσει το μικρόφωνο του μιλητή. Κύριε Γκέρεν, σας παρακαλούμε να ανάψετε το μικρόφωνο σας. Μα είναι αναμένο. Δεν, δεν σας ακούμε. Συνεχίστε. Ωραία, θα ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Σε αυτή τη συζήτηση θα τονίσουμε και πάλι πόσο σημαντικό ε, είναι να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση για όλα ε, τα δικαιώματα, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά. Ωραία, πολύ ωραία, δεν το αμφισβητώ αυτό. Αλλά ε, ε, υπάρχουν ναι, και κάποιες νόμιμες προσδοκίες. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεύτερης γενιάς δεν μπορούμε ε, να τα κατοχυρώσουμε, διότι τα αρχικά δικαιώματα της πρώτης γενιάς που προέρχονται από την Γαλλική Επανάσταση είναι ήδη κατοχυρωμένα, ενώ αυτό δεν συνέβαινε για τα κοινωνικά δικαιώματα. Ας μην μυρολατρούμε όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όργανα που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να κωδικοποιηθούν τα υπόλοιπα δικαιώματα όπως τα κοινωνικά παραδείγματο χάρη και μέσα από την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, βλέπουμε ότι δεν είναι όλα αυτά μια ψευδέση, μπορούν και να υλοποιηθούν. Ευχαριστούμε. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος ε, Μιγκάλσκι παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναγνωρίζω ότι δεν ήμουν θειασότης ε, της ε, θέσης ε, που προτείνεται, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι με τρία στοιχεία της παρέμβασης τελικά δηλώνω ικανοποιημένος. Ε, θα σας αποδώσω τα εύσημα. Ε, πρώτον, επιμείνατε στη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα φυσικά συμφωνούμε όπου και να είμαστε στη Λιβύη, στο Ιράν, σε οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να προστατεύουμε ε, πρωτίστως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, μιλήσατε για την καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας την πρόθεση της ανεξιθρησκείας. Πολύ ωραία. Ε, αλλά θα πρέπει να ακολουθούνται οι ιδέες και αποδράσεις. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι μετέχω στην αντιπροσωπεία για ε, συνεργασία με τη Λευκορωσία και χαιρετίζουμε την ευκαιρία που μας δίνεται να έχουμε μια ουσιαστική ανταλλαγή μέσα από την ίδρυση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επικροτούμε την απόφαση σας. Ευχαριστούμε για δύο λεπτά. Ο κύριος Μίτσελ τώρα παρακαλώ. President. Πρόεδρε, χαιρετίζω την ευκαιρία που μου προσφέρετε να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και ευθύ εξ αρχή θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την ενημέρωση εχθέ τη κυρία Υπατή Εκπροσώπου για θέματα που αφορούν στη Λιβύη. Έξι εκατομμύρια Εβραίοι δολοφονήθηκαν κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εδώ στην Ευρώπη. Ανάμεσα στους δύο πολέμους, τον πρώτο και τον δεύτερο, μιλάμε για 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους που δολοφονήθηκαν από όλα τα μέρη του κόσμου. Σύμφωνα με το περιοδικό Economist που δημοσιεύτηκε πρόσφατα ένα άρθρο, έχουμε 100 εκατομμύρια έλλειμμα γυναικών λόγω του ότι οι γυναίκες αυτές ε, χάνονται μόνο και μόνο γιατί είναι γυναίκες. Εχθές ήταν η, γυναίκα, η ημέρα των γυναικών, αυτό όμως το θέμα δεν ετέθη. Ε, πότε λοιπόν θα ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία έτσι ώστε να νιώθουμε σεβασμό και να μην επαναληφθεί αυτό που συνέβη κατά το πρώτο ήμιση του αιώνα. Εδώ το ίδιο το Κοινοβούλιο απαξιώθηκε. Καταψήφισε μία πρόταση να μην χρηματοδοτηθεί, να μην χρηματοδοτείται ο εξαναγκασμός σε άμπλωση. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι ε, συχάθηκα πλέον αυτή την πολιτική ορθότητα που δεν επιτρέπει τέτοιου είδου θέματα να συζητώνται στο Κοινοβούλιο με σεβασμό και ένα Κοινοβούλιο που να δέχεται και τι απόψει ε, τη άλλη πλευρά. Και ερωτώ την ύπατη εκπρόσωπο, αυτό το θέμα θα το θίξετε στα Ηνωμένα Έθνη. Και επιτρέψτε μου να σα πω τελειώνοντα ότι η στάση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ ε, στο ε, Στρασβούργο, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένες από τις αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου τις βρίσκω εντυπωσιακές. Μα πότε επιτέλους ε, θα μπορέσουμε να αποκαλύψουμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί εχθέ δεν εμφανίστηκε καμία γυναίκα που να πει ότι χάθηκαν αυτά τα 100 εκατομμύρια των γυναικών που δολοφονήθηκαν απλά και μόνο επειδή ήταν γυναίκες. Είναι λάθος που δεν φύγει το θέμα αυτό. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Μίτσελ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Ντεκάζερ, θέλει κάτι να σας επερωτήσω, να δηλαδή, υποδέχεστε την ερώτηση, ναι. Κύριε Ντεκάζερ. Αγαπητέ συνάδελφε, Κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα τη γιορτή τη γυναίκα, δεν θα πρόσεξα τότε στην ε, έκθεση τη κυρία Νεντέλτσεβα, που πρόκειται από τη δική πολιτική ομάδα, το θέμα τη ε, άμβλωση ήταν καθόλου ταμπού, διότι εμνημονεύθη, μνημονεύθη, ε, συζητήθη δημοκρατικά. Δεν πρόκειται περί ταμπού, πρόκειται περί τη δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω την θέση της κυρίας Ντεκάιζερ και τη σέβομαι Όσον αφορά στη δική μου την άποψη, πρέπει εδώ στο Κοινοβούλιο η μία πλευρά να ακούει την άλλη με σεβασμό και μετά να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Δεν άκουσα λοιπόν κανένα ούτε από τους σοσιαλιστές ούτε από τους φελεύθερους εδώ στο Κοινοβούλιο να φύγει το θέμα της άμβλωσης λόγω του φίλου Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταψήφισαν και ένα σχέδιο ψηφίσματος ε, να μην χρηματοδοτείται ο εξαναγκασμός σε άμβλωση. Αυτό λοιπόν είναι όνειδος, ντροπή για αυτούς που το έκαναν. Ας δείξουμε σεβασμό για τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Και για ένα λεπτό ζητεί το λόγο η κυρία Κοπά. Um, I think ο πρόεδρος. Νομίζω ότι η παρέμβασή σας προκάλεσε επερωτήσεις από τους άλλους αδέλφους. Αποδέχεστε, ναι. Έχετε το λόγο, κύριε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπάτη, εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίω και σέβομαι τις απόψεις του κυρίου Μίτσελ και θεωρώ ότι όπως και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο, και εγώ κατεδίκασα το ότι σε μια σειρά χωρών κοινωνιών στον κόσμο ε, το έμβριο, το θηλυκό ε, υφίσταται άμβλωση. Εξαναγκαστικό και άμβλωση, ανθρωποκτονία και. Όταν όμως το αναμειγνύουμε αυτό με το θέμα της αναπαραγωγής ελευθερίας, έτσι, το κουκουλώνεται, το υποβαθμίζεται, το κρύβεται. Το θέλει έμβριο. Να αναγνωρίσουμε το τι γίνεται και έτσι θα μπορέσουμε πιο εύκολα να συμφωνήσουμε. Μίτσελ, ευχαριστώ την αξιότιμη συνάδελφο κύριε Πρόεδρε. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να δίνουν περισσότερο σεβασμό ο ένα για τη γνώμη του άλλου. Και έτσι να προσπαθούμε να βρίσκουμε ένα κοινό παρονομαστή και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Οπότε παρακαλώ, α είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι. Εγώ βρίσκω πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να το χωνέψω το ότι το Κοινοβούλιο κατεψήφισε αυτή την τροπολογία για την χρηματοδότηση ή μη χρηματοδότηση ε, της ανθρωποκτονίας βάρος αυτών των εμβρίων. Ναι, και το πρόβλημά μου είναι το ότι όχι, όχι, δεν είμαι αναχρονιστής, δέχομαι να συζητήσω τα πάντα. Και τις απόψεις μου τις έχω τεκμηριωμένες και με, με, με χαρά μου τις με οποιονδήποτε και ευχαριστώ αυτούς που επερώτησαν. Καλά, α προχωρήσουμε, α αφήσουμε αυτό το θέμα, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα για 1,5 λεπτό θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κοπά. Κύριε Πρόεδρε, Λέδη Άστον, η Σύνοδο του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διεξάγεται φέτο στη σκιά των γεγονότων στη Βόρεια Αφρική και τον ευρύτερο αραβικό κόσμο, που έχουν πολλά να μα διδάξουν. Πρέπει ω Ευρώπη να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων. Είναι λοιπόν ευκαιρία να προχωρήσουμε σε ουσιαστική αξιολόγηση του Συμβουλίου, ώστε να βελτιώσει περαιτέρω τις μεθόδους εργασίας του αλλά και να υπογραμμίσουμε τη στήριξή μας στην ανεξαρτησία του και στο ρόλο του στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. σε αυτή την περίοδο των ιστορικών αλλαγών στη γειτονιά μας το μήνυμα της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. όμως παράλληλα οφείλουν και όλοι οι διεθνείς παράγοντες να εργαστούν για την εξάλληψη της πρακτικής των δύο μέτρων και δύο σταθμών στην επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβάλλεται να είμαστε συνεπείς και δίκαιοι όπως χαιρετίζουμε την πρόσφατη υιοθέτηση του ψηφίσματος που καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη λιβύη την ίδια σκληρή στάση πρέπει να κρατήσουμε και για την παράνομη συνέχιση του επικισμού στα κατεχόμενα της παλαιστίνης. ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Μίτσελ. Όταν μιλάμε για βασικά δικαιώματα, είτε αντρών είτε γυναικών, το σημαντικό είναι να μπορέσει να γεννηθεί κάποιος για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Πρώτη φορά ε, δέχονται κριτικές για τις διαδικασίες ε, που ακολουθούν στον αρμόδιο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών ε, και παρατηρούμε ότι υπάρχει μια διπλή ηθική, δύο μέτρα και δύο σταθμά διαπιστώνουμε πώς ε, μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση στην Λιβύη. Είδαμε την ε, στάση που τηρούν όλοι σε σχέση με το Ιράν. Ε, νομίζω ότι Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να εκδιωχθεί κάποιο από το Συμβούλιο και ξαναλέω εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και για την Λιβύη βλέπουμε επίσης πόσο διχασμένη είναι η διεθνής κοινότητα. Επίσης θα ήθελα να ε, ε, σχολιάσω το θέμα του Ισραήλ Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο ε, του Ισραήλ για την ε, δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, το Συμβούλιο αγνόησε τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών ε, στην προκειμένη περίπτωση. Άρα, έχει απολέσει και την αξιοπιστία του και πρέπει οπωσδήποτε ταχύτερο δυνατόν να θεωρήσει τον τρόπο εργασία του. Ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό, κύριο Όμπιολ. Πρώτα ευχαριστώ. Να μην επαναλάβω αυτά που προανέφεραν οι συνάδελφοι πάνω το είναι σημαντικά. Όμως θέλω να σας επισημάνω ότι σε αυτή την φάση των συνόδων του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι η κρίσιμη συγκυρία, η συμμετοχή της κυρίας ε, Άστον για μένα ήταν ε, καλά μαντάτα. Πρόκειται για να βγούμε προ τα εμπρό. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερη συνέπεια και προβάλλεται περισσότερο όσον αφορά τις ε, δράσεις της. Ε, έχουμε και θέσει σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα που μπορούν να κάνουν τα ανθρωπινά δικαιώματα και έτσι επίσης στο Συμβούλιο ε, συμπυγνωμίουμε κάποιες ε, συμμαχίες ε, αναγκαίες με άλλες ε, χώρες ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για διάφορα θέματα όπως το είπε και η κυρία Άστον θέματα που θα αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα Οπότε θα πρέπει κατά τον τρόπο για εμείς να διακηρύσουμε ότι δεν είναι το θέμα σχετικό. Είναι ε, κάτι, κάτι, κάτι απόλυτο. Είναι ε, αρχές με παγκόσμια ισχύ. Και επομένως θα πρέπει ακριβώς όπως καταφέραμε στο παρελθόν να καταργηθεί η δουλεία παγκοσμίω. Ελπίζω να καταφέρουμε η και ποινή παντού να καταργηθεί και να απαγορευτεί. Ευχαριστούμε κύριε Βιόρση, λέει ο Πρόεδρος. Για 1,5 λεπτό τώρα έχει το λόγο ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το απαραβίαστο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το σημαντικότερο σε μια κοινωνία. Ε, καθορίζει το επίπεδο των ε, δημοκρατικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα λάβει η χώρα στη Γενέβη πρέπει να έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Δηλαδή ε, η διακριτική μεταχείριση σε θέματα φύλου, ε, φυλής, ε, πολιτικού προσανατολισμού, η προστασία των μειονοτήτων και η προστασία των ευάλωτων ομάδων. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα και το Συμβούλιο λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα πολύ ευαίσθητο πλαίσιο. Αυτά που συμβαίνουν στη Βόρεια Αφρική και κυρίως στη Λιβύη είναι γνωστά σε όλους. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε μία μακρά συζήτηση και είχαμε παρεμβάσεις που τις εκτιμήσαμε Εκτιμήσαμε ιδιαίτερα εκτιμήσεις παρεμβάσεις εκ μέρους της κυρίας Άστον αλλά υπάρχει το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ακόμα ε, πιο ισχυρή ε, αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα, αλληλεγγύη. Αυτές θα πρέπει να είναι κατευθυντήρες γραμμές για συγκεκριμένες παρεμβάσεις χειρουργικές, διότι οι Μαροκινοί και οι Τινήσοι επιθυμούν να παραμείνουν εκεί που ζουν σήμερα. Και για να επιτευχθούν όλα αυτά πρέπει να ε, λειτουργήσουμε έγκαιρα. Θέλω λοιπόν να πω το εξή στην κυρία Άστον. Ε, καταγράψαμε αυτά που μας είπε πριν από λίγο και ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ουσιαστική διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τη θρησκεία. Οι πιο αιματηρές συγκρούσεις τους τον τελευταίο καιρό έγιναν ε, κατά των ε, χριστιανών ε, διότι υπήρχε, υπάρχει συγκεκριμένη χριστιανοφοβία. Ευχαριστούμε κύριε Κονέα. Τώρα πάμε στο ΚΑΤΣΔΙΑΕ. Πρώτη πρώτη έχει δει στο κύριε Νικολάε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Τι να σας πω, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον πρόκειται να αποτελέσει μια επιτυχία ή μια αποτυχία αυτή η σύνοδος. Όμως η συζήτηση εν λόγω θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει αποτελέσματα εκφραζομένη με μία ενιαία φωνή. Επομένως ε, είναι κακό ε, μήνυμα να το κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα που αρχίζει η Σύνοδος στη Γενέβη και στην Νέα και έτσι φανερώνεται το πόσο απουσία πολιτικής έχουμε. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε μιλώντας αποτελεσματικά και να δούμε κατά πόσον αυτό θα είναι ένας μηχανισμός παγκόσμιος για άμεση πρόληψη. Να μην περιοριστούμε σε απλή λήψη υπόψη των πεπραγμένων. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για πρόληψη στο μέλλον. Έτσι να έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Για ένα λεπτό, κύριε Στάνοκ. το γεγονό ότι η Λιβύη ήταν μέλος ε, του, ε, των ΗΕ, αυτό λέει πάρα πολλά. Ο Καντάφη για 42 χρόνια ήταν αρχηγός του κράτους και βλέπουμε τώρα τις συνέπειες της βίας και της τρομοκρατίας, τις οποίες βασιζόταν το καθεστώς. Υπάρχουν και άλλες καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από χώρες Κίνα, Κούβα, Σαουδική Αραβία, Ουγγάντα και αυτές είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί διώκουν τους ομοφιλόφιλους. Στο Ιράν δεν υπάρχει επιτροπή ισότητας των γυναικών ε, δαπανώνται ε, πάρα πολλά χρήματα ε, για το Ισραήλ, αλλά θεωρώ ότι όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, πράγματι ας μη γελιόμεθα υπάρχουν αντιφάσεις δηλαδή μη δημοκρατικά καθεστώτα που είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δοκιμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Στίβενς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Άστον. Βαρόνι Άστον, δεν απαντήσατε στον κύριο Ζάρατελ στην προηγούμενη συζήτηση για το Ιράν, για τον Καμπάσρα. Ε, ε, οι 3.400 αυτοί άνθρωποι υφίστανται βασανιστήρια, παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. 1,2 δις δίνουμε για την ανοικοδόμηση του Ιράκ και παρόλα αυτά κάθε φορά που ψηφίζουμε εδώ μία πρόταση στο Κοινοβούλιο, κάθε φορά που κάνουμε μία γραπτή δήλωση και εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία, μας αγνοεί ε, η Ιρακινή κυβέρνηση ε, και Ξέρετε ότι ψυχολογικά βασανίζουν αυτούς τους ανθρώπους στον ε, καταβλισμό. Έχουν τα μεγάφωνα που όλη την ημέρα ε, ε, προωθούν την προπαγάνδα του καθεστώτος εδώ και ένα χρόνο. Ε, Επίση, το νοσοκομείο για όσους έχουν τραυματιστεί και όσους πάσχουν από καρκινό δεν λειτουργεί. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, να τους πούμε. Δεν θα σας δώσουμε άλλα χρήματα αν δεν αλλάξετε ρότα. Ευχαριστούμε κύριε Στίβενσον. Για ένα λεπτό η κυρία Τότς. Uh, um, Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ήπατη εκπρόσωπο το εξή, Βλέποντας όλα αυτά τα γεγονότα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και βλέποντας ε, επίσης ε, ότι υπάρχει γενικότερα μία αγωνία όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ύπατη εκπρόσωπος ε, θα στηρίξει εκείνους στον Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν συγγενείς ε, οι οποίοι δολοφονήθηκαν ε, λόγω της ε, έκρηξης βομβών ή από τα πυροβόλα όπλα του Καντάφη και των απαντών του. Και κυρία Άστον, θα στηρίξετε το νέο καθεστώς που θα προκύψει από τη σύγκρουση στη Λιβύη. Ευχαριστώ κύριε Ντότς. Τελευταίος να δώσω το λάβει το λόγο για το ΚΑΤΣΤΙΑ γιατί ήδη έχουν περάσει τα χρονικά όρια. Για ένα λεπτό κύριο Σαραφράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα πλαίσια της συζήτησής μας που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε σχέση με την έκθεση που προηγουμένως συζητήσαμε κύριε Άστον, έχω την εξή ερώτηση. Θεωρείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα όσα γίνονται σε αυτές τις χώρες της Βορείου Αφρικής και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι τώρα τόσο εύστοχο να στείλουμε στο Ιράν μια αντιπροσωπεία, να ανοίξουμε μάλλον συγγνώμη ένα γραφείο και μια αντιπροσωπεία τη Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Σαραφρανικά. Και τώρα το λόγο έχει η Πάτη εκπρόσωπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δείξατε πάρα πολλά θέματα. Εγώ το πρώτο που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για την ενέργεια και το πάθος με το οποίο ε, μίλησαν σε αυτή τη συζήτηση. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που δημοσιεύτηκε η έκθεση κυρίας Ανρίκεν για την ε, εξέλιξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ε, και βέβαια έκτοτε θεσπίστηκαν και άλλα ψηφίσματα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά της και για τη δουλειά της ε, ε, βοήθησε έτσι ώστε ε, να οικοδομηθεί και η δική μας υπηρεσία. Χαίρομαι που η κυρία Χάουταλα θα μεταβεί στην συνέλευση του Συμβουλίου. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι θα συμμετάσχει σε αυτή τη συνέλευση γιατί έχει πολύ καλές και εμπεριστατωμένες γνώσεις η κυρία Χάουταλα. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι ε, πιέσαμε να υπάρξει αναθεώρηση και βεβαίως ε, η αναθεώρηση δεν είναι όσο καλή θα θέλαμε αλλά βλέπουμε τώρα ότι ε, θα υπάρξει η μεταφορά στη Νέα Υόρκη θα συνεχιστούν εκεί οι εργασίες οι βουλευτές που συνεργάζονται μαζί μας μπορούν να επιφέρουν σημαντική ε, αλλαγές. Εγώ είμαι, νιώθω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η κυρία Χάουτρα θα ε, οθήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, που μου ετέθησαν. Ο κ. Χάουτς είπε όσον αφορά το DRC πράγματι Θεωρώ ότι συμφωνούμε και πράγματι πρέπει να υπάρξει ένα ψήφισμα. Στο Πακιστάν ε, στις 5 Μαρτίου είχαμε συγκεκριμένη ε, παρέμβαση για το άρθρο 30. Ε, Στα άλλα μέλη που μίλησαν για την ελευθερία των θρησκευτικών πεπιθήσεων, σας πω καταρχήν ότι Πράγματι ε, μιλάμε για ε, φρικαλές τραγωδίες ε, χριστιανών ανά τον κόσμο, σε πολλά μέρη του κόσμου. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το δικαίωμα της θρησκευτική ελευθερίας ε, είναι κατοχυρωμένο και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε ε, να εκφράζουμε τις απόψεις μας, να καταδικάζουμε την τρομοκρατία ή επιθέσεις σε θρησκευτικέ κοινότητες συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανών. Η δική μου ομάδα, οι συνεργάτες ε, θα συναντηθούν με τους ευρωβουλευτές για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε Αναφέρομαι στο τι μπορεί να κάνει και συγκεκριμένα ε, το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, κατά τα άλλα, νομίζω ότι έχουμε περίπου 3.400 Έχουμε εβδομαδιαία επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη που επισκέπτονται τους καταβλισμούς των προσφύγων έτσι ώστε να καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες. Ε, πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει στην Καπάσρα και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, και διαφορετικές απόψεις επί του θέματος. Όμως ο κύριος Ευρωβουλευτής έχει απόλυτα δίκιο ότι το σημαντικότερο είναι να διασφαλίσουμε την ε, ακαιρεότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Επειδή σας είπα ενημερώνομαι κάθε εβδομάδα πράγματι προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατά τα άλλα, να σα πω ότι συμφωνώ επίση ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι να στείλουμε μια ισχυρή αντιπροσωπεία στη Γενέβη. Η κυρία Χάουταλα το έθιξε αυτό επίση. Μόλι ορίσαμε νέο επικεφαλή ε, τη αντιπροσωπεία. Εγώ ε, όταν πήγα στη Γενέβη ε, μίλησα με την αντιπροσωπεία. Ξέρετε, χωρίσαμε στα δύο την αντιπροσωπεία. Η μία θα ασχολείται με θέματα του ΠΟΕ και το άλλο ημισή θα ασχοληθεί περισσότερο με τους οργανισμούς ε, των Ηνωμένων Αθνών. Επίσης, στις συζητήσεις που διεξήγαγα είπα ότι πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο παραγωγικά ε, το πώς λειτουργούμε στη Γενέβη. Πρέπει να έχουμε συμμαχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μπορούμε να μιλάμε με εταίρους ανά τον κόσμο, να κάνουμε κοινή μας υπόθεση ορισμένα σημαντικά θέματα που απασχολούν όλους μας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε επικεντρώσουμε σε αυτό κατά τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και μήνες. Και να σας πω επίσης ότι αυτά ε, που είπε ο κ. Σαλαβράκος με εντυπωσίασαν πάρα πολύ όταν είπε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τρόπος ζωής. Και έχει δίκιο σε αυτό. Εγώ ε, είπα πολύ απλά ότι ε, για να νιώθει κανείς ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει κανείς να είναι ανθρώπινος είναι πολύ σημαντικό ό,τι και αν κάνουμε να μην ξεχνάμε αυτή την τόσο σημαντική αρχή. Ε, ε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, υπάρχουν πολλά θέματα επί των οποίων μπορούμε να διαφωνούμε, όμως ε, το να μπορούμε να συζητάμε για τα θέματα αυτά και να τα βάζουμε στο επίκεντρο της σκέψης μας, νομίζω αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Και τέλος θέλω να πω ότι δεν έχω αποφασίσει κατά πόσον θα υπάρχει υπάρξει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν. Ε, θα σας ενημερώσω εν το χρόνο και εντωμεταξύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και να ξέρετε ότι προσπαθούμε το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να το κάνουμε όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται και μόνο αυτό θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπροσωπούνται σε θέματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο αποτελεσματικότερα γίνεται. Κύριε Σαλαφράγκα, ζητείτε το λόγο. Δεν κατάλαβα καλά τι απήντησε η κυρία Άστον. Γιατί νομίζω ότι είπε ότι αυτό το οποίο ρώτησα εγώ όσον αφορά το κατά πόσο εύστοχο είναι να έχουμε αντιπροσωπεία στο Ιράν ε, αν αυτό θα αναβάλλεται ε, ή δεν απάντησε καθόλου. Γιατί ε, σύμφωνα με τη διατύπωση των όσων άκουσα δεν, δεν, δεν πήρα απάντηση. Κυρία Άστον. Βεβαίω, κύριε Σαλαφράγκα, προσπαθούσα να πω ότι έχουμε δύο χωριστά θέματα. Πρώτα-πρώτα το θέμα των πόρων, μοιραία. Και το δεύτερο, ότι απαιτείται να ληφθεί η σχετική απόφαση κατόπιν προτάσεώ μου για την αντιπροσωπεία. Και βεβαίω, πρώτη αυτόν ζητήσει σε Κομισιόν, Συμβούλιο και σε εσά. Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα. Η δέσμευσή μου για το Ιράν γνωρίζετε αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τα πυρηνικά. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κλείνει το μικρόφωνο. Έχω λάβει έξι αιτήματα σχετικά με προτάσεις ψηφίσματος και αύριο το μεσημέρι θα γίνει η ψηφοφορία.